την προτείνει ε, ώστε να ισχύει η εντολή από 25 Νοεμβρίου του 2015. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Με βάση το άρθρο 105 παράγραφος 6 ο πρόεδρος της διάσκεψης ε, ο Πρόεδρος των επιτροπών με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς δύο συστάσεις από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου Προϋπολογισμών σχετικά με την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Δεν τάσσονται κατά, οι προτάσεις ισχύουν αν δεν ταχθούν 40 μέλη κατά μέσα σε 24 ώρες. Αλλιώς θα, οι συστάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία και υπάρχει και